Ολοκληρώθηκαν έτσι οι παρεμβάσεις του ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 150. Ακολουθεί τώρα η παρουσίαση του κυρίου Ρούμπιχ για τις μικρομεσαίε επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα, ο οποίος έχει το λόγο για 4 λεπτά. Mm. Κύριε Ρούμπιχ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην ε, Ολομελία είναι μεγάλο το ενδιαφέρον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πάντα χαίρομαι για το ότι αναγνωρίζετε το οικονομικό δυναμικό τους και ξέρουμε πως 58% των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη δημιουργείται από εταιρείες οι οποίες ε, υπάρχουν πέντε χρόνια ή λιγότερα. Και αυτό δεν σχετίζεται με την ηλικία της εταιρείας αλλά με την ηλικία του ιδρυτή. Και βεβαίω πρέπει να τονιστεί και η κουλτούρα του να είναι κανείς επιχειρηματίας στην εκπαίδευση, γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Ήδη από τον υπηαγωγείο πρέπει να μάθουμε τα παιδιά να είναι ανεξάρτητα και πολλά παιδιά και πολλοί άνθρωποι στην Ευρώπη θέλουν να είναι ανεξάρτητοι, γι' αυτό νομίζω πως είναι σημαντικό να δούμε και τους ε, business angels, τους ε, χρηματοδότες αυτούς, αλλά βεβαίως να δούμε πώς αποτελεί και μια σημαντική ευκαιρία για γυναίκες, νέους και μετανάστες. Βλέπουμε λοιπόν πως ε, η Κομισιόν έχει ανέλαβει εδώ πέρα μια σημαντική πρωτοβουλία. Δυστυχώς στην Ευρώπη δεν είμαστε πάρα πολύ επιτυχημένοι με την βιομηχανική πολιτική μας. Έχουμε μείωση κατά 10% από το 2008 θεωρώ πως θα ήταν σημαντικό εδώ πέρα να κάνουμε τα, τα λεγόμενα τεστ μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις ε, διάφορες χώρες. Εδώ πέρα η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν γίνονται δηλαδή σωστά αυτά τα τεστ και να υπάρξουν μετά θετικές προτάσεις για το πώς μπορούμε να κάνουμε κάποιες απλοποιήσεις. Και ένα πόρταλ επίσης πολύγλωσσο θα ήταν σημαντικό εάν δείτε το τι γίνεται, τι εξάγεται και τι εισάγεται από άλλες χώρες, ποια είναι τα προβλήματα, οι ευκαιρίες και στον τομέα ειδικά των εξαγωγών για μικρές επιχειρήσεις ειδικά με το ίντερνετ, με τα διεθνή συστήματα πληρωμών, με τις ε, υπηρεσίες αποστολών ε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τις τεχνολογίες επικοινωνίας υπάρχουν πάρα πολλές νέες ευκαιρίες και εδώ πέρα επίσης είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε με τους ανθρώπους και επίσης σημαντικό είναι το πρόγραμμα Εράσμους για τους νέους επιχειρηματίες και πρέπει να ενισχυθεί πάρα πολύ στην περίοδο μέχρι το 2020. Το βλέπουμε αυτό ειδικά στις χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα ε, στον τομέα της συνοχής. Είναι πάρα πολύ θετική η αντιμετώπιση αυτού του προγράμματος και θα μπορούσε να είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Mundus να επεκταθεί παγκοσμίω έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή με τους προμηθευτές τους, με τους πελάτες τους, ε, είναι επιχειρηματίες, να μάθουν νέες αγορές για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά του. Εδώ πέρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί βεβαίω και το Enterprise Europe Network γιατί υπάρχει ήδη αρκετή πείρα εκεί πέρα και είναι ένα τομέα ο οποίο μπορεί να επεκταθεί νομίζω παγκοσμίω για να έχουμε μεγαλύτερες επιτυχίες. Αλλά η ανταγωνιστικότητα σημαίνει πως πρέπει να σταματήσει και η γραφειοκρατία, η μείωση του διοικητικού άχθους. Στόχος θα ήταν μέχρι το 2015 να έχουμε μια μείωση κατά 25% του διοικητικού άχθους. Και εδώ πέρα λοιπόν θα μπορούσε η Επιτροπή των Περιφερειών να κάνει κάτι προς αυτή η κατεύθυνση. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τα της φορολόγησης και το πώς θα γίνεται να μεταφερθεί μια επιχείρηση από τον άνθρωπο στον άλλον. Σας ευχαριστώ. Παίρναμε, λοιπόν κατευθείαν στη διαδικασία Catch the Eye. Να δώσω τον λόγο στην κυρία Ματσέη Κουκουβίτση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαίρω τον δόκτωρα Παλ Ρούμπιχ. Έχει κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά μαζί με άλλους σε καιρό κρίσης. Η δουλειά αυτή είναι σημαντική έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε απαντήσεις για αυτό το οποίο μας περιμένουν αύριο. Αυτή είναι η σημαντικότερη πρόκληση. Τι μας περιμένει αύριο και στην έκθεση αυτή νομίζω πως υπάρχουν απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα. Υποστηρίζω. Τον κύριο Ρούμπιχη όταν μιλάει πως ε, για το ότι πρέπει να υπάρξει ήδη από τον υπηαγωγείο εκπαίδευση για την ε, επιχειρηματικότητα και για την τόλμη, γιατί χωρίς αυτή δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα. Και θα πρέπει τα ευρωπαϊκά δίκτυα επιχειρηματιών να έρχονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μας λένε συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είχαν, πόσες startups προέκυψαν παραδείγματο χάρη από κάθε δίκτυο. Σας ευχαριστώ κυρία Ματσικούκοβιτς. Κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όλοι σε όλα τα κόμματα θέλουμε οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ένα καλό περιβάλλον εργασίας. Αυξάνουν τις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προωθούν την ανάπτυξη και είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και υγιείς και ικανοποιημένους εργαζόμενους. Η έκθεση Ρούμπιχ δίνει εδώ πέρα ένα λανθασμένο μήνυμα. Γιατί ε, λέει πως ε, τα της υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι γραφειοκρατία. Προδιαγραφές ασφαλείας και ελάχιστες προδιαγραφές δεν είναι διοικητικό βάρος. Λέτε πως ε, τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να επιβάλλουν υψηλότερες προδιαγραφές από αυτές τις οποίες επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα επειδή όλα αυτά είναι ελάχιστες προδιαγραφές, το να ε, επιβάλλονται αυστηρότερες προδιαγραφές από τα κράτη-μέλη επιτρέπεται πάντα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βέρτμαν. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 23 εκατομμύρια μικρομεσαίες επιχειρήσεις, απασχολούν 75 εκατομμύρια ανθρώπους, μιλάμε για ένα ποσοστό που είναι πάνω από το μισό των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί σε καιρούς κρίσεις αποτελούν ένα μήνυμα αποφασιστικότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία και οπωσδήποτε ένας κινητήρας μπορεί να συνεισφέρει και συνεισφέρει στην ανάπτυξη και στην αηφορία. Και τέλος να ευχαριστήσω τον κύριο Ρίμπη για τη λεπτομερή του έκθεση. Σας ευχαριστώ κυρία Βέρτμαν. Κυρία Τσούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε ίσως να συμφωνήσουμε με την έκθεση αυτή. Αναφέρεται σε μια σειρά από μέτρα για τη διάδοση πληροφοριών κλπ. Η έκθεση όμως αυτή δεν επικεντρώνεται στα βασικά προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στην Πορτογαλία οι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν καθημερινά λόγω της πολιτικής λιτότητας που έχει επιβάλει στην υπάκουη κυβέρνησή μας η Τρόικα. Οι πολιτικές αυτές οδηγούν σε μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης και την απώλεια ε, αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. Όλα αυτά οδηγούν στη μείωση της οικονομίας μας. Αυτές οι πολιτικές λιτότητας, αν συνεχίσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως στις χώρες μας, θα δυσκολέψουν πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητά μας και οι επιχειρήσεις στη χώρα μου δεν θα μπορέσουν να αναπτυχθούν. Κάνω έκκληση για αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη θα μείνει νεκρό γράμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι και πόρο απέχει από την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος κύριος Μικολάση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ευκαιρίες που έχουν θα πρέπει να είναι η σημερινή, το σημερινό μας θέμα. Γιατί αν θέλουμε να πούμε ότι η πολιτική συνοχής, να μιλάμε για πολιτική συνοχή σημαίνει ότι πρέπει να στηρίζουμε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και την ανταγωνιστικότητά τους. Πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ε, πολλά κερδίσει από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία και αυτό έχει βοηθήσει την απασχόληση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε τις περιβαλλοντικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες στο χώρο της γεωργίας ή της βιολογικής γεωργίας Ιδίως αν, θέλουμε να λυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα στις διάφορες περιοχές. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα διορθωτικά ταμεία θα πρέπει και αυτά να έχουν επαρκείς πόρους για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μικολάσικ. Και τώρα η συνάδελφος Ανδρές Πάρια. Παρίγια. Παρίγια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το 75% λέει ο εισηγητής ε, των θέσεων εργασίας ε, ε, είναι, το, το, το, το δημιουργούν οι ΜΜΕ οι οποίες όμως δεν εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς και δεν αναπτύσσονται πέρα από τα σύνορά τους. Τι να κάνουμε ρωτάει ο εισηγητής για να μειώσουμε το γραφειοκρατικό άγχος να αυξήσουμε την διεθνοποίηση, να μπορέσουμε να έχουμε ένα, ένα Erasmus των επιχειρήσεων για το προσωπικό. Χρειάζεται όμως και πρόσβαση στη χρηματοδότηση και δεν κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται εν ώψη του 2020 να ενισχύσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στις ΜΜΕ, να μπορούν οι ΜΜΕ να έχουν πρόσβαση στα δάνεια που σήμερα δεν έχουν. Πρέπει να τις διευκολύνουμε στα δάνεια γιατί εκεί ε, ε, έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία. Ζητούμε ως θεμελιώδες στοιχείο να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα δάνεια οι επιχειρήσεις, οι ΜΜΕ για να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ κυρία Παρίγια, ο κύριος Βίνκλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Ριμπιχή για την έκθεση αυτή ως συζητητής για την γνωμοδότηση της ΙΝΤΑ ε, συνεργάστηκα και εγώ μαζί του τονίστηκε ήδη πώ μεταξύ των στόχων της έκθεσης είναι να ενισχυθούν οι συνθήκες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς και να αντιμετωπίσει κάποια εμπόδια ε, που εμποδίζουν αυτή τη στιγμή τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν στο διεθνές ε, εμπόριο. Θεωρώ λοιπόν πως αυτές οι πληροφορίες οι οποίες θα δίνουν και οι δημόσιες αρχές και ενώσεις μία είναι πάρα πολύ σημαντικές όσον αφορά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τρίτες αγορές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα νέα κράτη-μέλη είναι σε μειονεκτική θέση οπότε πρέπει να έχουν ειδικέ πληροφορίες με τρόπο πιο προσβάσιμο. Τέλος, η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ακολουθεί η κυρία Φλασίκο Βαμπένοβα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολούν 75 εκατομμύρια ανθρώπους και 75% όλων των θέσεων εργασίας και έχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Τα δεδομένα δείχνουν πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο κινητήρας της ευρωπαϊκής οικονομίας να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να επιτύχουν την ενσωμάτωση, αλλά έχουν πολλά διοικητικά βάρη, γραφειοκρατία, εμπόδια στην ε, συστασική ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υπάρχουν πάρα πολλά, δεν έχουν πρόσβαση σε δάνεια, υπάρχουν προβλήματα στην διαχείριση των διαφορετικών ταμείων και συχνά η ενίσχυση η οποία υπάρχει δεν τους φτάνει. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση, ο κύριος Κέλλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτή τη φάση ασχολούμαστε με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρούμπιχ για αυτό που επεσήμανε και να ενθαρρύνω την υλοποίηση της έκθεσης αυτής. Κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο κύριος Ρούμπι είχε αναφέρει και σημασία της παιδείας. Το έχουμε συχνά παραλείψει. Πηγαίνω συχνά στο σχολείο και ρωτάω τα παιδιά τι θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν. Πολλά παιδιά μου έχουν πει ότι θέλουν να είναι επιχειρηματίε, να έχουν δική του επιχείρηση. Και έχει δίκιο ο κύριο Ρούμπικ. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τον υπηαγωγείο να δημιουργήσουμε αυτό το ενδιαφέρον, αυτή την κουλτούρα. Επίση, αυτό το θέμα της γραφειοκρατίας που λέει είναι σημαντικό και κυρίως η δοκιμασία για η δοκιμή των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις και είναι ε, μεγάλες οι δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα πρέπει να τις ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν είδα την κυρία Τσικάου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Mulțumesc, domnule președinte. Οι επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττονται από την οικονομική κρίση επειδή η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι δύσκολη το 85% των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2010 ως το 2012 δημιουργήθηκαν από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι η βιομηχανία παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. 25% των θέσεων εργασίας στο ιδιωτικό τομέα προέρχονται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να τις στηρίξουμε και σε τοπικό και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην ενιαία αγορά και στις αγορές των τρίτων χωρών. Πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στις πληροφορίες, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας να προστατεύονται. Χρειάζεται καλύτερη πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορικής. Χαίρομαι, το ε, χαιρετίζω το νέο πρόγραμμα COSME που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ελπίζω ότι όλα τα ευρωπαϊκά μέσα να τις διευκολύνουν, κυρίως αυτές, αυτά που επιτρέπουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία και τη ΔΙΑΕ. Και τώρα θα ακούσουμε τον Επίτροπο τον κύριο Πίμπαλξ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, θα ήθελε η Κομισιόν να ευχαριστήσει τον κύριο Ρουμπί και τους ευρωβουλευτές οι οποίοι συνεισέφεραν στην έκθεση το οποίο δείχνει το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Κομισιόν καλωσορίζει την ε, στήριξη στις ε, δράσεις που ανακοινώθηκαν ε, για την διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βιομηχανική πολιτική και την απορρίθμιση. έχετε δίκιο, αντιπροσωπεύουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις γύρω στα 2 τρίτα των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα και 58% της προσθέμενης αξίας και 85% των νέων θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια. Όμως έχουν επηρεαστεί κατά πολύ από την κρίση και βεβαίως πρέπει να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις. Η Κομισιόν μπορεί να σας διαβεβαιώσει πως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική θα εστιαστεί στην προώθηση των δραστηριοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω πολλών προγραμμάτων, μέσω της απλοποίησης ε, διαδικασιών και της δημιουργίας μόνο απευθυντικών υπηρεσιών. Αλλά βεβαίως και μέσω της παροχής υπηρεσιών που απευθύνονται ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το COSME, Επίση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Η έκθεση του κυρίου Ρουμπίχ μιλάει για μια στρατηγική διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η Κομισιόν το υποστηρίζει. Αυτή τη στιγμή μόνο 13% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξάγουν εκτός της Ένωσης και όλοι γνωρίζουμε πού βρίσκονται οι ευκαιρίες για ανάπτυξη σε οικονομίες που βρισκονται οι ευκαιρίε για αναπτυξη σε οικονομίε που αναπτυσσονται γρηγορα στην Ασία, Νότιο Αφρική και ε, στην Νότιο Αμερική και ο ΣΑ υπολογίζεται πως, υπολογίζει πως η περισσότερη ανάπτυξη μετά το 2012 θα λάβει χώρα εκτός της Ένωσης. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα κενά της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο εξωτερικό. Τα αποτελέσματά μας θα παρουσιαστούν τον Δεκέμβριο του χρόνου. Θα έχουμε συγκεκριμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που ε, αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όμως σας διαβεβαιώ πώς θα συνεχίσουμε με τις επιτυχημένες πρωτοβουλίες που έχουμε ήδη όπως το πρόγραμμα Enterprise Europe την υπηρεσία επαφή με την ε, Κίνα και βεβαίως τα κέντρα τρίτων χωρών. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω εδώ πέρα και το τις αποστολές για την ανάπτυξη του ε, Επιτρόπου του κ. Ταγιάννη που ήταν το 2012 στο Μεξικό, Κολομβία, Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες και είχαμε θετικές αντιδράσεις καθώς και πολιτικές συμφωνίες σε διάφορους τομείς όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η βιομηχανική συνεργασία. Όσον αφορά την μείωση του διοικητικού βάρους, αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί όλους, η Κομισιόν ενισχύει αυτή τη στιγμή το τεστ μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά όπως ξέρετε εξακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβαρύνονται από διάφορους κανονισμούς. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή σε στενή συνεργασία με μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούμε να βρούμε τις 10 πιο επιβαρυντικές νομοθεσίες και ξεκινάμε ε, Βεβαίω μια δημόσια διαβούλευση η οποία συνεχίζεται μέχρι τα Χριστούγεννα. Δεν έχουμε καιρό να χάσουμε και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα μας επιτρέψει να δούμε τα προβλήματα. Θα ελέγξουμε την προβληματική αυτή νομοθεσία και θα δούμε που υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξει ένα πιο ελαφρύ καθεστώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πάντα βέβαια λαμβάνουν υπόψη τις πτυχέ της υγείας και της ασφάλειας αλλά πλέον και ο προπολογισμό Ένωση θα δώσει στοχευμένη στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα COSME θα καλύψει δράσεις ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως τη βελτίωση πρόσβασης σε χρηματοδότηση και το δίκτυο Enterprise Europe. Επίσης, σκοπεύουμε να βελτιώσουμε την βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την πρόσβαση σε αγορές εντός και εκτός της Ένωσης. Όλα αυτά προτεραιότητες που αναφέρονται στην έκθεσή σας κύριε Ρουμπίχ. Επίσης το κόσμο θα ενισχύσει το Εράσμους για επιχειρηματίες που ανέφερε ο κύριος Ρουμπίχ. Οπότε το κόσμο είναι ένα πρόγραμμα που θα ενισχύσει τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Σε αυτούς τους καιρούς λιτότητες είναι σημαντικό το ότι αυξάνεται ο προπολογισμό αυτού του προγράμματο. Συνοψίζοντα, ο πρόεδρο τη Κομισιόν, ο κ. Μπαρόζο, έχει τονίσει επανειλημμένω πω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι βασική προτεραιότητα τη θητεία του και σα διαβεβαιώ πω ε, σκοπεύει να το εφαρμόσει αυτό χρησιμοποιώντα όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε εδώ η συζήτηση. Ψηφοφορία αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Θα ακολουθεί τώρα η έκθεση Oyuland ε, για περιορισμούς θεώρησης ε, διαβατηρίων για Ρώσους αξιωματούχους που είχαν εμπλακεί στην υπόθεση Σεργέη Μανίτσι. Τον λόγο έχει η κυρία Όγιουλαντ.